Ladies and gentlemen, I'm going to um, start the meeting. τη συνεδρίαση κυρίες και κύριοι, λέει η πρόεδρο αν είναι δυνατόν και πρώτα πρώτα να κλείσουμε την ημερησία διάταξη. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό μεταδίδεται στο ίντερνετ, η συνεδρίασή μας δηλαδή, και όλα τα έγγραφα για τη συνεδρίαση υπάρχουν στην εφαρμογή η meeting εγκρίνεται το κείμενο των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση. Και αν δεν υπάρχουν στάδια θα έρθουν εγκριθμένα πρακτικά στο τέλος της συνεδρίασης. Σε αυτό το σημείο συνέδριο γίνεται μια ενημέρωση με του τριμμένου διαλόγου και σα υπενθυμίζω ότι θα υπήρξε ενημέρωση, αλλά όχι για τέτοιες συνεδριάσεις, αλλά σε άλλες συνεδριάσεις όπου κάποιο συνάδελφος από την Επιτροπή έχει πάει για να μας εκπροσωπήσει. Γι' αυτό και θέλω να υπάρξει μέσα στη διάταξη το, το σημείο για την ενημέρωση και επίσης μια ομάδα εργασίας για το copyright, τα το copyright. Ντάνιελ, μπορείς να μας ενημερώσει για το τι έγινε στην τελευταία συνεδρίαση που είχες παραστεί και τι έγινε και με την ομάδα εργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα και το copyright. Α, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, μετάδοση της Γερμανίας σε όλο το κτίριο. Ή τέλος πάντων κάποιες, κάποιες ε, καμπίνες ακούγονται, κάποιες όχι. Τα γερμανικά ακούγονται, ρωτάει ο πρόεδρος. Τσεχικά. Αλλά βλέπω ότι όλα τα άλλα δεν λειτουργούν. Άρα θα πρέπει η τέλο πάντων, παντων καποιες καποιες καμπινες ακουγονται καποιες οχι τα γερμανικα ακουγονται ρωταει ο προεδρος τσεχικα αλλα βλεπω οτι ολα τα αλλα δεν λειτουργουν αρα θα πρεπει η τεχνικη να ασχοληθούν με το πρόβλημα. Οπότε, εμείς ας συνεχίσουμε με τον Ντένιελ Ντάλτον που να μας κάνει αυτή την ενημέρωση για το τι έγινε ε, στην συνεδρίαση για το copyright. Ε, αυτό θα μας το πει στα αγγλικά, τα ακούσουμε στα αγγλικά και θα έχουμε μετάφραση αργότερα. Let's start with Daniel Επομένως, ξεκινούμε με τον ε, Ντάνιελ και... και όταν υπάρξει μετάφραση, για να θέλει να μας τα ξαναπεί. Οπότε, Ντάνιελ, για να δούμε, θα δούμε θα γίνει το επόμενο σημείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ ότι είπα, αν χρειαστεί να τα πω ξανά. Και το πρώτο που έχω να σας πω για τη συνεδρίαση εκείνη είναι ότι η ΙΜΚΟ εκπροσωπήθηκε πάρα πολύ καλά. Ήταν η Τζούλια εκεί από την Επιτροπή την νομική και η Σαμπίνη Φερχάγεν. Οπότε βλέπει την αντιμετώπιση του copyright και των προηγούμενων δικαιωμάτων. Σε δύο μετά έγινε η συνεδρίαση. Πρώτα-πρώτα είχαμε τον Πράτσης ε, ο οποίος παρέστηκε γενικώ ήταν μια κάπως βαρετή συζήτηση όπως αυτές που κάνουμε εμείς εδώ δεν πρόκειψε τίποτα καινούριο ε, τίποτα για το νόμιμο για τις εξαιρέσεις και αυτά που Τζο επίσης τα, έχουμε ξανασυζητήσει αλλά θα δούμε τι επιτροπή τι θα πει γιατί θα καταβληθεί προσπάθεια να δούμε πώς όλα αυτά θα επιληθούν. Και το δεύτερο μέρος της συζήτησης συζητήθηκαν και τα γεωσκόπη δεδομένα και μετά συζητήσαμε για τα δεδομένα, την άντληση των δεδομένων όσον αφορά την παιδεία, την επιστήμη και την υγεία. Μας τα εξήγησαν, ε, μας προβλημάτισαν και τι να πούμε μετά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και εντυπωσιαστήκαμε από το τι δυνατότητες προσφέρονται όσον αφορά αυτό το πεδίο, αυτό το τομέα της άντλησης των δεδομένων. Η πρόεδρο σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλους τους συνάδελφους της Επιτροπής οι οποίοι μας ε, εκπροσώπησαν σε αυτές τις συναντήσεις. Τώρα αφορά το κανάλι 6 ή από το κανάλι 6 μέχρι το 12 λειτουργεί κανονικά. Όμως η διερμηνία από τα άλλα κανάλια δεν λειτουργεί. Πρόκειται να λάβει μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν υπάρχει διερμηνία. Um, Δεν ξέρω. Κύριε Σφαμπ. Τι λέει κύριε Σφαμπ. Δεν λέει. Δεν ξέρω. Μήπως. Να, κοιτάξτε, το πρώτο θέμα είναι για το Νεόχτ και για την Ελβετία, οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε τελείο υπόψη σε αυτό. Ε, θα έχουμε τουλάχιστον ε, διερμηνία προ τα γερμανικά και προ τα γαλλικά. Δεν ξέρω τώρα Μήπω γίνεται οι να αλλάξουν θέσεις. Αλλά βέβαια τι θα γίνει και με τους άλλου, με τι άλλες γλώσσε. Και μόνο να σε ρωτήσω, μήπως οι άλλες γλώσσες δεν χρειάζονται σήμερα, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί μπορεί κάποιο που μιλάει αυτή τη γλώσσα που θέλουμε να κόψουμε ούτω ή να θέλει να ακούσει τον ομιλητή. Άρα νομίζω ότι το πιο να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Και. Όχι, τεταρτάκι. Και θα ξαναρχίσουμε στι 4.30. So the update, ladies and gentlemen, is that the electricity... Κυρίες και κύριοι, μόλις αποκαταστάθηκε η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα και γίνεται ένα reboot τώρα στι συσκευές. Οπότε προτείνω να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και θα ε, στις και μισή ξαναρχίζουμε, χωρίς κανένα πρόβλημα.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 Α, εντάξει, έχουμε προς τα γαλλικά διερμηνία. Ωραία. Και γερμανικά. Σας μπέρδεψα. Με ακούτε. Έχουμε γερμανικά. Γερμανία προς τα γερμανικά. Στο κανάλι παριθμών ένα είναι τα γερμανικά. Και δουλεύει. Ναι. Ωραία. And no waves coming from translation booth. Thank you very much. Okay, we're going to move straight to... Οπότε, κατευθείαν να το προχωράμε και πάμε στην έκθεση της πρωτοβουλίας του Ανδρέας Φβάμπ και αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και οπότε θα προσπαθήσουμε τώρα να καλύψουν το χρόνο μας ένα 25 λεπτό και 4 παρα 5 έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα. Αντρέα, δεν Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Πρέπει να ομολογήσω ε, ότι αισθάνομαι κάπω άβολα που κάνατε τόση φασαρία για αυτή την έκθεση. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας. Για δεύτερη φορά τη συζητά η Επιτροπή μα. Ε, συμφωνία με τι χώρε ΕΖΕΣ ε, και την ε, Ελβετία, ΕΟΧ δηλαδή, είναι μια γερή συμφωνία που λειτουργεί καλά και παρά ε, τις πολλές εσωτερικές εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις χώρες ΕΟΧ και στην Ελβετία από την άλλη, έχει αποδειχθεί στην πράξη ως εργαλείο μέσω επέκτασης της ενιαίας αγοράς σε τρίτες χώρες. Μπορεί να πούμε ότι σήμερα δεν θα προσφερόταν μια τέτοια συμφωνία στο εσωτερικό της Ευρώπης γιατί τους δίνει μια σειρά από προνόμια που κανονικά πρέπει να είναι αποκλειστικότητα το μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και ο συνάδελφος Ράφαλ Τρασκόφσκι που είχε κάνει την έκθεση πριν από πέντε χρόνια έχει σημειώσει ότι είναι μια γερή βάση στην οποία μπορούσαμε να οικοδομήσουμε. Ταυτόχρονα όμως και επίσης ισχύει το εξής. Ε, και οι χώρες ΕΖΕ, ΕΟΧ πρέπει να κάνουν περισσότερα, όπως και τα κράτη-μέλη της Ένωσης άλλωστε, για να ε, ε, υιοθετούν, να υλοποιούν, να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τη λειτουργία του κοινοτικού δικαίου στο δικό τους χώρο, στην ένωμη τάξη. Γιατί υπάρχει μια αρχή για την παρακολούθηση ο επόπτης της ΕΦΤΑ, της ΕΖΕΣ, που έβγαλε τώρα την 35η έκθεση και στο βαθμολόγιο λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 2% η επίδοση στο βαθμολόγιο και στην Ελβετία πώς γίνεται. Από τη μια η νομοθεσία τους αναγνωρίζεται ως σχετική με τον ΕΟΧ και από την άλλη ε, μεταφέρεται στο εθνικό τους δίκαιο. Και ε, ήδη από το πρώτο βήμα υπάρχει καθυστέρηση, οπότε καταλαβαίνετε ότι και στο δεύτερο υπάρχουν δυσκολίες και καθόλου ε, ευκαταφρόνητες. Και στην ευρωπαϊκή ε, εσωτερική αγορά, αν θέλουμε να κάνουμε βήματα πρόοδου στην ε, διακυβέρνηση, αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις χώρες ΕΖΕΣ και ΟΧ. Από την τελευταία θητεία με εισηγητή του συνάδελφου Τρασκόφσκι, τι έχει προκύψει. Οι Ελβετοί και Ελβετές στις 9 Φεβρουαρίου του 2014 κάνανε ένα δημοψήφισμα και Ξέρετε ότι υπάρχει ένα σημείο της συμφωνίας των χωρών μας με την Ελβετική Συνομοσπονδία ε, και αμφισβήτησαν κάποια βασικά στοιχεία και στο μεταξύ το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος ε, θα ε, γίνει, είναι καθοδόν για να γίνει εθνικό δίκαιο. Ξέρετε ότι και εγώ και πολλοί το βλέπουμε αυτό επικριτικά γιατί τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εσωτερική αγορά ε, συνοδεύονται και ισότιμα με κάποιες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες ΕΖΕΣ και ΕΟΧ και καλούνται να τις εφαρμόσουν και σήμερα και στο μέλλον. Οπότε θα κυριαρχήσει στην έκθεση αυτή αυτό το στοιχείο, έχετε την έκθεση όλοι στα χέρια σας. 7 Μαΐου θα κάνουμε και ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας για να εμβαθύνουμε και ε, θα κυριαρχήσει το ζήτημα αυτό του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, από τη μία, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι ώστε η υλοποίηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως έχει να εξασφαλίζεται και στις χώρες ΕΖΕΣ και ΟΧ, ένα αυτό. Και δεύτερον, ποια είναι η πολιτική απάντηση στην ε, πρωτοβουλία κατά της μαζικής μετανάστευσης στην Ελβετία που κινδυνεύει να ανατρέψει τις διμερείς συμφωνίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία ε, ή τουλάχιστον να τις αμφισβητήσει. Ξέρω ότι η γνωμοδοτή Επιτροπή Απασχόλησης, δεν έχει μεταφραστεί αυτή η γνωμοδότηση, ε, αν κατάλαβα καλά θα γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή Εξωτερικών, ΑΦΕΤ, και οι δύο γνωμοδοτήσεις είναι για μένα σημαντικές και θα τις λάβω υπόψη φυσικά στην επόμενη δουλειά. Υπήρξαν και μερικά σημεία που για λόγους έτσι, χώρου ε, δεν τα έβαλα στην έκθεση μου, αλλά θα συμπληρωθούν με τροπολογίες ε, έφθετο ε, χρόνο. Περιμένω να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τους και όλες Ευχαριστώ. Μαρία Γραπίνη. Γραπίνη. Έχετε το λίγο, το λόγο για, για την Σοσιαλδημοκράτες κύριε Γραπίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Ανδρέας με συντομία μας παρουσίασε την έκθεσή του και εγώ συμφωνώ ότι το πρόβλημα με την Ελβετία ακόμη δεν έχει διευθετηθεί. Φυσικά και το δημοψήφισμα είναι έκφραση ε, δημοκρατίας, αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να λάβουμε όλε τι ευθύνε μα για τη συνεργασία μεταξύ μα. Η έκθεση είναι πάρα πολύ εύστοχη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα όσα γνωμοδότησαν και οι δύο επιτροπέ. Υπάρχουν ακόμη όμω κάποια προβλήματα. Προβλήματα που αφορούν τη συνεργασία. Πρόκειται για εγκάρσια οριζόντια ζητήματα, πρόκειται για πάνω από 100 ε, συμφωνίες κλαδικές. Επομένως, θα ήταν προτιμότερο εάν μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας γινόταν να συναυθεί μια συμφωνία. Να συμμετάσχετε στον ΙΟΧ η Ελβετία και όχι μόνο σε αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα της ελεύθερης διακίνησης προσώπων. Εδώ αναφέρεται και το πώς θα επεκταθεί αυτό στην Κροατία. Οπότε βλέπουμε ότι οι σχέσεις με την Ελβετία επιδέχονται βελτίωση. Σε θα συζητήσουμε και άλλο και στις πολιτικές ομάδες και να δούμε πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση των σχέσεων. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον συγητή, λέει κυρία Τρεμπέσιος, ε, για την εκτενή του παρουσίαση. Ένα μεγάλο τμήμα των συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ελβετίας είναι προϊόν διμερούς διαπραγμάτευσης και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Όπως είπε και ο εισηγητής, ε, διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην εφαρμογή και καλό θα ήταν να ε, μπορούσαμε να σημειώσουμε βήματα πρόοδου. Το πιο δύσκολο στοιχείο των διαπραγματεύσεων είναι τι γίνεται με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ε, της 9 Φεβρουαρίου 2014 κατά της μαζικής μετανάστευσης. Η ομάδα μου είναι υπέρ μιας ε, αποκεντρωμένης Ευρώπης με επικορικότητα και το κόμμα μου ε, υποστηρίζει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ελβετία. Θα πρέπει η λαϊκή βούληση να γίνεται συμβαστή οπωσδήποτε. Και εδώ δύο θέματα θα πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, η δυσλειτουργούσα ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε τι γίνεται στη Μεσόγειο και υφίσταται τι συνέπειε και η ε, Ελβετία. Και θα θέλαμε να την καλέσουμε να βοηθήσει την ε, Ελβετία και να συνεχίζει να προστατεύει τα εξωτερικά ε, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωση, και μάλιστα να εντείνει τι προσπάθειε Λόγω των οικονομικών κρίσεων στη Νότια Ευρώπη είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε υποστήριξη από την Ελβετία. Και σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ήταν καλύτερα τα πράγματα, ήταν μικρότερη επιβάνηση για την Ελβετία, αλλά λόγω της κρίσης, κατά κύριο λόγο, ο κόσμος πηγαίνει στις περιφέρειες όπου η ε, οικονομία λειτουργεί καλά και δημιουργούν και κοινωνικά προβλήματα στους ε, αυτόχθονες μεταξύ άλλων αυξάνονται τα ενίκια Φερρυπίν ως συνέπεια. Έχει αποτύχει η νομισματική πολιτική και δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Και η κατάσταση που επικρατεί τώρα δεν πρέπει να καταλογιστεί στην πολιτική της Ελβετίας που απέτυχε, αλλά στην πολιτική της Ευρωζώνης που απέτυχε. Η Ελβετία είναι μια χώρα κυρίαρχη και κάνει πολιτική για τον ίδιο της το λαό και αυτό αξίζει σεβασμού. Εμείς είμαστε λοιπόν πρόθυμοι να συμφωνήσουμε με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, προσβλέπουμε και ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία μαζί τους και θέλουμε να βελτιωθεί και η οικονομική συνεργασία, ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας και της δυνατότητας αποθήκευσης αυτής. Ε, επειδή είναι δύσκολη να γίνει αυτή η ενεργειακή αλλαγή στη Γερμανία ε, ε, είναι κρίσιμη και πολύτιμη συνεισφορά της Ελβετία, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Γερμανίας και σε ό,τι αφορά την αυτόματη ε, πληροφόρηση για θέματα καταπολέμησης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το θέμα στο TTIP, να δούμε τι γίνεται με τα συστήματα επίλυσης ε, διαφορών και προστασίας του επενδυτή. Ε, πάντως, νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε και διμερώς με τον εισηγητή και είμαι αισιόδοξη ότι θα καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ola Tunas is the ALDE shadow, but Robert Rochefort is going to speak for ALDE. Merci, Présidente. Euh, Madame Tornaes s'excuse. Ο κ. Ροσφορή, η κυρία Τμός ε, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα το απόγευμα, ζητάει συγγνώμη, έχει συντάξει ε, ένα σημείωμα το οποίο και θα σας διαβάσω. Η Συμφωνία ΕΟΧ είναι μια επιτυχία ιστορική σημασία, χάρη στην οποία μπορούν να εισέρχονται στην κοινή αγορά χώρε, έχοντα μια πρόσβαση σε μια αγορά 500 ε, εκατομμυρίων καταναλωτών. Όμω, ε, ε, είναι προϊόν διαπραγματεύση ιστορική και με τι εξελίξει τη συνθήκη τη Λισαβόνα θα πρέπει να επανεξετάσουμε την λειτουργία του ΕΟΧ για να αποκομίσουμε τα μέγιστα ωφέλη. Οι διοικήσεις καθυστερήσεις στην εθνική μεταφορά κάποιων νομικών πράξεων όντως οφείλονται εν μέρη σε αναγκαίες προσαρμογές. Όμως οι καθυστερήσεις ε, αυτές πλήττουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου στην ε, ενιαία αγορά και θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης, ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι ακρογωνιός λήθος τη νέα αγορά. Ε, και γι' αυτό η λαϊκιστική εκστρατεία που έγινε το ε, Φεβρουάριο του 2014 με εκείνη τη δημοσκόπηση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι βασική εγγύηση για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να επικρατήσει συνοχή και με κοινωνικο-οικονομικά βιώσιμο τρόπο να ρυθμίσει το πρόβλημα πρόβλημα της μαζικής μετανάστασης. Ε, η συμφωνή ε, με το περιεχόμενο της έκθεσης του κυρίου Σφάμπ και ε, μην ξεχνάμε ότι έπεται και μια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Κάθριν Στάινερ. Ένα λεπτάκι. Υπάρχει κάποιος από τους πρασίνους από το, την Κούερ. Α, Πασκάλ, ζητώ συγγνώμη, δεν ήσουν στη λίστα μου. Βίκη, για τους πράσινους ε, θα τα πω γρήγορα διότι δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω τη δουλειά που έκανε ο Ανδρέας. Ε, ιδιαίτερα μας ικανοποιεί ότι επιμένει στη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της νομοθεσίας ε, στις χώρες ΕΖΕΣ. Δεν υπάρχει ε, καμία φοβερή δυσκολία. Συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις που έκανε. Φυσικά, από πλευράς της Ισλανδίας υπάρχει ένα πολιτικό έλλειμμα για το οποίο λυπούμαστε και επίσης είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό μη ενσωμάτωσης για τη μεταναστευτική πολιτική της Ελβαϊτίας θα συμφωνήσουμε με τον εισηγητή Μία τροπολογία νομίζω μόνο θα καταθέσουμε που σχετίζεται με το θέμα της εφορολογικής σύγκλησης. Ε, με την Ελβετία δεν νομίζω να ξαφνιάζουμε κανέναν. Ε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν άκουσα καλά στο σημείο ένα, μήπως είναι και πρόβλημα μετάφρασης. Είναι λίγο αμφίσιμη η δήλωση του Αντρέα, αλλά δεν νομίζω να ήθελε να πει αυτό, ότι ε, είναι βασική κινητήριο δίωμα τη οικονομία η συμφωνία και ο στόχο είναι να επεκταθεί η ενιαία αγορά σε τρίτε χώρε. Δεν νομίζω να είναι αυτό ο στόχο μα, ότι θέλουμε να εξάγουμε αυτό το μοντέλο. Μάλλον ε, είναι θέμα διατύπωση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα η Κάθριν Στέλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις. Αυτή η έκθεση του κυρίου Σφάμπα είναι μια καλή επισκόπηση και περιγραφή της ε, κατάστασης. Είναι σημαντικό, όπως ε, κάνατε και εσείς, να ε, κάνουμε την διαφοροποίηση ανάμεσα στο, στην ενία αγορά και την συμφωνία ΕΟΧ, τη διαφορά που υπάρχει κυρίως στα σημεία 3 και 6. Βλέπουμε τα προβλήματα με τις χώρες ΕΖΕΣ, η Ισλανδία παραδείγματος χάρη, ε, στο Free Tech ε, τα είπαμε σε πρόσφατα στην Νορβηγία. Ε, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και θα πρέπει να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο το ζήτημα. Τώρα για την Ελβετία το σημείο 14 της έκθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως, όπως και είπαν κάποιοι συνάδελφοι, πως πρόκειται για μια απευθεία επίθεση, κατά μέτωπο επίθεση κατά των Γερμανών και των Ιταλών που δουλεύουν στην Ελβετία. Ε, χρειάζεται παρακολούθηση. Στις 12 Ιουνίου στη συνεδρίαση με την ε, μεικτή αντιπροσωπεία έχει, θα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το ζήτημα, πρέπει να το αναφέρετε το θέμα της παρακολούθησης. Επίσης ε, ε, φαντάζεστε ότι στις 7 Μαΐου δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί λόγω των εκλογών στη χώρα μας. Επίσης ε, περιμένουμε και την ε, δημόσια ακρόαση για αυτό το ζήτημα και ελπίζω να μοιραστείτε μαζί μας τα πορίσματα. Προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστούμε. Ωραία. Θέλω και εγώ να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθεί η Επιτροπή τι γίνεται με την νομοθεσία αφού την εγκρίνουμε. Μεταφέρεται ή δεν μεταφέρεται στην Εθνική Νομοθεσία και εφαρμόζεται ή όχι. Ε, για τη νομοθεσία που σχετίζεται με την ενιαία αγορά είναι ένα πάγιο ζήτημα αυτό, η μη μεταφορά δηλαδή στην εθνική νομοθεσία ε, και άρα ξεκάθαρα κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το κατανοήσουμε. Εάν κάποιες ομάδες χωρών φαίνεται να μην μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τα νομοθετήματα, τότε θα πρέπει να ε, δούμε για ποιο λόγο. Επίσης, να πω ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάποιους τομείς της ενιαίας αγοράς και ζητώ και πάλι από τη γραμματεία ε, ζήτησα μάλλον το κεφάλαιο από την γραμματεία μου πει ποιοι είναι οι τομεί αρμοδιότητά μα. Ε, ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, τεχνικά πρότυπα, ελευθερία εγκατάσταση, ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, λειτουργία ε, της εσωτερικής αγοράς για όλους τους προαναφερθέντες τομείς. Όμως ο συντονισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπών δεν είναι της αρμοδιότητός μας. Ε, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να στρέψουμε την προσοχή μας στους τομείς που ε, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Αποσχόλησης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ε, διότι δεν, για άλλους φακέλους όταν ε, πάω και διεκδικώ την αρμοδιότητά μας ε, σε κάποιον τομέα μου λένε ότι μπαίνω στα χωράφια τους. Ε, ξέρω ότι είναι ένα φορτισμένο συναισθηματικά ζήτημα και θέλετε να το συζητήσετε, αλλά προσεκτικά μην πατήσουμε τον κάλο των άλλων επιτροπών γιατί, γιατί αυτό υπονομεύει και το δικό μου το ρόλο όταν εγώ προσπαθώ να υπερασπιστώ του τομείς όπου ε, έχουμε και την μεγαλύτερη δύναμη λοιπόν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Είναι δική μας δουλειά ε, να παρακολουθούμε αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Ε, προσοχή όμως για το, στο παράρτημα 7 του ιστορικού κανονισμού όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας στον τομέα της νέας αγοράς. Βοηθήστε με να μην υπερβαίνω τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ο Γιαννούκα Γρήγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Εργάζομαι στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Αλλά θα μιλήσω για λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε για το σχέδιο τη ε, έκθεση. μέσα στο ίδιο μήκο κύματο. Ακριβώ όπω και τα συμβασμάτα του Συμβουλίου για μια επέκταση και ομοιογενή ε, επέκταση της ε, αγοράς όπως οφασίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου. Επομένως, πρόθυμα θα συνεργαστούμε. Η Πρόεδρος. Κύριε Σιγητά, θέλω να παρέμβετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφέρω τα εξή τρία στο τέλος της συνεδρίασης πριν πάμε στο επόμενο θέμα λόγω χρονικής πίεσης. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους ε, και τη Γραμματεία φυσικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα είπανε. Ελπίζω τους επόμενους μήνες να έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε και να ε, καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή. Δεύτερον, χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Στάιλε, ο Πασκάλ Ντουιρόν και εσύ αγαπητή Βίκη, αγαπητέ Πρόεδρε, Εθίξατε το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίηση της ε, κοινοτικής Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για την έκθεση αυτή είναι βασικά ε, κεντρική ιδέα και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Σας είπα ε, στην 35η ενημέρωση η ημερωση η γραμματεια ΕΖΕΣ το εντοπίζει αυτό, ότι επιβραδύνεται η εφαρμογή στις χώρες ΕΖΕΣ και ΟΧ. Και εμείς έχουμε ε, αρμοδιότητα για την ενιαία αγορά στα κράτη-μέλη βάσει του κανονισμού και θα πρέπει να παρακολουθούμε και την εφαρμογή, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι στις τρίτες χώρες. Ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα για την Ελβετία. Βέβαια, είναι ειδική περίπτωση σε αυτή την υπόθεση γιατί δεν ανήκει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αλλά ε, ε, είναι πάρα πολύ προχωρημένη ολοκλήρωση. Και εσείς, Πρόεδρε, μιλάτε και είπατε ότι δεν πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, αλλά η ίδια σας η συνάδελφος της πολιτικής σας ομάδα, η κυρία Τρεπέζιους, το έθεσε. Στην Ελβετία το θέμα δεν είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά των εργαζομένων και των υπηρεσιών. Και υπάρχουν και κάποιες παρεξηγήσεις, γιατί αν δεν υπήρχαν θέσεις Εργασία στην, Ευρω... Ελβετία, τότε δεν θα έβαζαν και μετανάστες. Αυτό είναι η όλη παρεξήγηση. Δημιουργείται η ε- εντύπωση, χωρίς να υπάρχει κανένα ε, στοιχείο στον κανονισμό του Κοινοβουλίου, ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα προσφύγων και ένα πρόβλημα ελεύθερης κυκλοφορίας. Μα είναι ένα πρόβλημα ε, αγορά εργασία. Επειδή σφίζει λοιπόν η αγορά εργασία στην Ελβετία, πηγαίνει ο κόσμος εκεί και εργάζεται. Εάν δεν διατίθεται αυτέ τι θέσει, δεν θα πηγαίνει ο κόσμο. Παρακαλώ λοιπόν να τηρήσουμε αυστηρά τον κανονισμό μα. Περί τίνο πρόκειται και τι μα ενδιαφέρει εμά η ενιαία αγορά και να εξασφαλίσουμε τι ελεύθερε κυκλοφορίε στην ενιαία αγορά, στην εσωτερική, όχι μόνο στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε τρίτε χώρε που έχουν πολύ ε, υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης, όπως είπε και ο Πασκάλ Ντυρό. Γιατί αποφάσισαν από μόνοι τους ότι ε, δεν θέλουν να συμμετάσχουν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να μην είναι κράτη-μέλη δηλαδή, αλλά να έχουν τα οικονομικά οφέλη. Οπότε θα πρέπει να εφαρμόζουν την νομοθεσία που κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για λογαριασμό τους και όλα τα υπόλοιπα θα ήταν ε, αντίθετα με τη συνθήκη. Και παρακαλώ να τα πούμε αυτά στου φίλου και γείτονε μα ΕΟΧ και ΕΖΕΣ και στην ίδια ε, την Ελβετία ότι τα μέσα αυτά που αυξάνουν την ευημερία ε, θα λειτουργήσουν μόνο εφόσον όλοι ε, τηρούν τα όσα έχουν συνυπογράψει. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. So, um, we are going to have a... Επομένως, στις 7 Πέμπτου πρόκειται να γίνει μια ακρόαση, η τροπολογία μέχρι τις 12 Μαΐου και θα συζητήσουμε τροπολογίες 22 και 23 Ιουνίου. Και 15 Εβδόμου οι συμφεστικές τροπολογίες θα ψηφίσουμε δε στις 16 Ιουλίου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. eating up time. We can do a quick change to the next. Ελπίζουμε το χαμένο εδώ για να δούμε το επόμενο θέμα. Αλλάζουμε θέσεις, μια που είμαι εγώ εισηγήτρια. Okay, we're moving on to the reports and person. Ford. Μέσα ατομικής προστασίας. Η συγκέντρια είναι Vicky Ford. Mm. Είστε έτοιμοι, μάλιστα. Έχουν γίνει οι συζητήσει ανταλλαγή απόψεων και με ε, ηλεκτρονική επικοινωνία, με τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Σα ευχαριστούμε που μου είπατε σε ποια σημεία μπορούμε να πετύχουμε κάποιο συμβασμό. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε δύο σημεία. Πρώτα-πρώτα το πεδίο εφαρμογή και κατά δεύτερο όσον αφορά την απροστεμένη διαδικασία για την ανανέωση τη εξέταση τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε κάποιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ο κανονισμός δεν περιέχει κάποια διερεύνηση για διευκρίνηση. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το ΕΛΚ, θέλουμε κάτι να υπάρξει όσον αφορά την άριστη πρακτική και θα πρέπει ο κατασκευαστή να μπορεί να χρησιμοποιήσει την προστατευμένη διαδικασία για να νιώσει το πιστοποιητικό και κάθε πενταετία να μην ξεκινάει από το Α. Οπότε, αν υπάρχει δηλαδή μια αλλαγή, να πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία. Ένα δεύτερο θέμα αφορά το πεδίο εφαρμογής, όπως θα θυμάστε, το κείμενο της Επιτροπής προέβλεπε το να διευρυνθεί αυτό το πεδίο εφαρμογής για κάποια οικιακά προϊόντα. Κάποια τα οποία δεν είχαν υπαρχθεί σε κάποια ρύθμιση προηγουμένως. Και υπήρχαν κάποιες προτάσεις για συμβαστικές τροπολογίες σε σχέση με το τι προβλεπόταν πριν 25 χρόνια. Ε, μεταξύ αυτού και του τι προβλέπεται να γίνει τώρα. Κάποια παραδοσιακά προϊόντα, είπαμε ότι να μην καλυφθούν τα οικιακά προϊόντα. Ας πούμε τα γάντια για την ε, λάντζα και ε, κάποιες φωσφορίζουσες ταινίες πάνω στα ρούχα αυτό επομένως να μην καλύπτεται. Οπότε γίνει και τα προϊόντα προστασίας κατά της θερμότητος. Εάν αυτά τα προϊόντα το ισχυρίζονται αυτό, δηλαδή ότι το προϊόν σας προστατεύει κατά της θερμότητος, ε, κάποια γάντια, τότε θα πρέπει να καλύπτονται. Εάν δεν ε, το ισχυρίζεται αυτό ο κατασκευαστής, τότε δεν θα καλύπτονται από το νομοθέτημα. ούτως ώστε να υπάρχει η προστασία εκεί που χρειάζεται. Περισσότερες πολιτικές ομάδες έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους. Δεν έχουμε όμως ε, εδώ του, τον σκιώδη συγκητή από τους σοσιαλιστές για να συζητήσει. Okay. So the first shadow Ο πρώτος γεωσηγητής. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Αριμόντ. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία, ε, για τη συμβαστική πρόταση αυτή. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ πάρα πολύ ε, με τις προτάσεις σας, γιατί έχετε συμπεριλάβει και πολλές δικές μας. Έχω μερικές σύντομες παρατηρήσεις όμως. Στην συμβαστική πρόταση υπαριθμών 1, αυτό είναι ένα μικρό τεχνικό σχόλιο, λέγει ότι καλύπτεται από αυτή την οδηγία. Μα δεν είναι οδηγία, είναι κανονισμός, ξέρετε. Μήπως να αλλάξει αυτό ε, ε, που έχουμε παραβλέψει. Και στην τελευταία πρόταση, σε αυτή τη συμβαστική πάντα, που παραπέμπει στο ε, παράρτημα 1 της οδηγίας 89 κάθετος 686 πρέπει να, κατα... σας πω ότι δεν έχω κατανοήσει τις προθέσεις μας αρχικά. Εγώ θεωρούσα ότι όλα αυτά τα πράγματα που είναι ήδη εκτός, του πεδίου εφαρμογή ε, ρυθμίζονται εκ των υστέρων ε, με κατεξουδότηση πράξης. Έτσι θεωρούσα ότι μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή. Και εδώ στα πλαίσια της Επιτροπής μας κανονικά το έχουμε συζητήσει Και τώρα το πεδίο εφαρμογής ορίζεται πάρα πολύ συγκεκριμένα και πάρα πολύ στενά, που εμένα με βρίσκει υπέρ. Αλλά τώρα δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ πώς να το ερμηνεύσω αυτό, πώς να το εκλάβω, γιατί δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Και σας ερωτώ λοιπόν, αν μπορούσε η συγγήτρια να μας τα εξηγήσει σύντομα αυτά. Επίσης χαίρομαι που αρκετά νωρίς λέει το κείμενο ότι το πεδίο εφαρμογή ορίζεται βάσει του παραρτήματος 1. Καλό είναι αυτό. Και εξασφαλίζει και κάποια ασφάλεια δικαίου ακριβώς, γιατί υπάρχει συναντήληψη. Συμφωνώ και με την συμβαστική πρόταση για τις ανακλαστικές επιφάνειες. Και ένα σημείο τριβής τώρα δεν είναι μόνο το πεδίο εφαρμογή, αλλά και η διάρκεια. Διότι εμείς ξαναγράψαμε το κείμενο από την αρχή και πάνω κάτω τα λέει και η σχετική τροπολογία, η δικιά μας. Εγώ προβληματίστηκα ε, πώς θα πρέπει να οριστεί η διάρκεια στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται πενταετία. Αλλά χωρίς απλουστευμένη διαδικασία και αν δεν αλλάξει τίποτα. Η δική μου πρόταση κανονικά θα ήταν να... Να είναι αυτό ελάχιστη διάρκεια. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής, μάλλον η πρόταση της ηγήτριας και η συμβαστική είναι να είναι το μέγιστο αυτό. Βέβαια παραμένει για μένα το ερώτημα τι γίνεται με προϊόντα που δεν έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής Μήπως ανοίγουμε διάπλατα τις σύρες για το παρατηρητήριο ή για διάφορες αρχές ε, που μελετούν τα προϊόντα για να μειώσουν ε, τις διάρκειες και τις προθεσμίες. Οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να ελέγχονται συχνά και να επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες πιστοποίησης, πράγμα που θα επιβαρύνει προφανώς και διοικητικά την επιχείρηση που τα παράγει και τη διαδικασία πιστοποίησης και για εκείνου που κάνουν την πιστοποίηση και πληρώνονται γι' αυτό, του συμφέρει να είναι μικρότερη διάρκεια για να ανανεώνεται αυτή η διαδικασία. Οπότε με προβληματίζει αυτό. Υπάρχουν όμως τώρα μέσα ατομική προστασίας που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, που δεν ε, είναι πενταετία. Και αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Η μέγιστη διάρκεια ζωής ε, δεν με ενθουσιάζει, αλλά μπορώ να τη δεχτώ. Θα δω με κάποιο τρόπο να κάνω μια τροπολογία για να μην επιβαρύνουμε πολύ διοικητικά τις εταιρείε ε, στα μέσα ατομικής προστασίας. Δηλαδή να μην λήγουν μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια οι άδειε και να πρέπει να πιστοποιούνται από την αρχή τα προϊόντα. Κατά τα άλλα συμφωνώ με το συμβιβασμό, μπορούμε να το δεχτούμε και ευχαριστώ τους συναδέλφους και την εισηγήτρια φυσικά την κυρία Φόρτ. Ευχαριστούμε κυρία Άριμοντ. Για να συγχωρευτούμε ότι δεν υπάρχει άλλος από εδώ. Για να μιλήσει για άλλη πολιτική ομάδα. Ο κύριο ε, ο κύριος ευχαριστούμε για τα τόσα ενδιαφέροντα τα οποία έχετε επεξεργαστεί και για τη συνεργασία σας. Εμείς ως η ομάδα των ε, σκιωδών εισηγητών ε, υποστηρίζουμε αυτές τις συμβαστικές που νομίζω ότι καλύπτουν τη γνώμη όλων μας. Και όσον αφορά τις πρώτες που είναι για το παιδί θα πρέπει να πούμε ότι να καλυφθεί ό,τι χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό λέμε λίγα λόγια. Δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια της λογικής. Και ε, ό,τι χρησιμοποιούμε καθημερινά, άπαξ και ο κατασκευαστής δεν ε, ε, ισχυρίζεται κάτι ιδιαίτερο στον αυτή την προστασία, δεν θα πρέπει εμεί να μπερδεύουμε τα πράγματα, οπότε συμφωνούμε επί της ουσία αλλά όχι βέβαια 100% με όλα όσα είπε ε, το ΕΛΚ, οπότε θα πρέπει να να, να, μην, να μην καλύψουμε 100% των, ε, των προϊόντων ό,τι έχει σχέση δηλαδή με την ασφάλεια. Άρα επομένω να κάνουμε αυτό το συμβασμό στον φρόντο πεδίο εφαρμογή και αυτό το οποίο κάναμε είναι ικανοποιητικό. Τώρα αυτό το οποίο μα είπε η Βίκη πριν από λίγο όσον αφορά αυτά τα διακοσμητικά ε, στοιχεία τα οποία όμως είναι φωσφορίζοντα, αυτά μπορούν να ε, εξαιρεθούν από σχεδόν υπάρχει προστατευτική λειτουργία η οποία να ε, προτείνεται ως ισχυρισμός του κατασκευαστή. Επομένως το κείμενο θα διευκολύνει τα πράγματα. Γιατί πολλές φορές δεν είναι τόσο σίγουρα τα πράγματα και διαχωριστική γραμμή μεταξύ του τι είναι μόδα και του τι είναι χρηστικό α το πούμε αντικείμενο δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Οπότε όταν πρόκειται για μόδα ή για διακόσμηση τότε είναι θεμητή αυτή η ρύθμιση. Άπαξ και δεν έχουμε σχετικό ισχυρισμό του κατασκευαστή. Ας εξαιρείτε το προϊόν τώρα όσον αφορά τη διάρκεια ε, της πιστοποίησης. Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα για την πιστοποίηση. Γιατί καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο καθένας εξημών, αλλά θεωρώ ότι αυτή η συμβαστική τροπολογία είναι αξιόλογη. Άκουσα τι είπε και το και οπότε θεωρώ ότι το αντίβαρο ας πούμε του ότι προτείνουμε μία πάρα πολύ απλή διαδικασία είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η πενταετία ως μέγιστο όριο και όχι ως ελάχιστο. Κάτι σαν ασφαλιστική δικλίδα. Ότι δηλαδή ακριβώς εν ώψη της επιστήμης, αν δεν υπάρχει κάτι το καινούριο, εάν η βιομηχανία δεν ε, αλλάζει το προϊόν, ε, τότε η απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται είναι πάρα πολύ εύκολη, πραγματικά. Και δεν νομίζω εδώ πέρα υπάρχει ενός εκτροπής για κάποιους ενδιάμεσους οι οποίοι πρόκειται να επιβαρύνουν περισσότερο όπως ελέγχθη και λοιπά και λοιπά όσον αφορά τον καταναλωτή. Επομένως νομίζω ότι προς τα εκεί προσανατολίζεται ο συμβασμός και επομένως είναι εύστοχος. Μία ερωτησούλα έχω τώρα για την δίκη, για την εισηγήτρια. Εγώ κατέβασα μια τροπολογία που αφορά την προστασία των μοτοσυκλετιστών αφορά και εμένα τον ίδιο. Από τα 14 καβάλα μοτοσυκλέτα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσει το κείμενο σαν αφορά τα προστατευτικά ρούχα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο παράγων ασφάλεια στα ρούχα αυτά. μαζί δηλαδή, αυτά που είναι ενσωματωμένα στο, στο, στο, στο ρούχο σε σχέση με τη χρήση του. Γιατί όταν κάνουμε την αξιολόγηση του προστατευτικού κινητού στοιχείου ε, ε; αυτό, όμως δεν συμβάλλει αναγκαστικά στην ασφάλεια. Όμως σε συνδυασμό με τη, με την μπλούζα, ε, ανάλογα το πώς φρενάρουμε, πώς τρίβουμε, ε, αλλάζει το θέμα του πόσο προστατεύει. Άρα έτσι θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση. Σφαιρικά, συνολικά και έτσι να αξιολογούμε αυτά τα ρούχα. Ελπίζω να συμβάλλει. Επίσης, Μπράβο για άλλη μια φορά για την έκθεση και όλα θα πάνε καλά με το κείμενο. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Ρασφόρ για να δούμε. Είναι κανείς άλλος εδώ. Όχι, α, δεν υπάρχει άλλος και ο ηγητής. Α, ο κύριος Ντυρέ. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα άκουσα από όσα μας, είπε στην εισήγησή της η και με τον Ρομπέρ συμφωνώ και εγώ από τα 14 καβόλα μου το συγκλέτω οπότε δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω πάντοτε θα πρέπει να προσέξουμε να είναι ουσιαστική και όχι θεωρητική η ασφάλεια νομίζω ότι με αυτή την αποθεμένη διαδικασία επανεξέτασης έχουμε τώρα μια πρόβλεψη, μια ρύθμιση πάρα πολύ ισορροπημένη. Οπότε, να μην το παραψάχνουμε περισσότερο. Ήδη ήταν δύσκολο να καταλήξουμε κάπου για το πεδίο εφαρμογή. Ήδη είναι αρκετά προληπτική ρύθμιση. Τώρα το θέμα είναι να έχουμε ασφάλεια δικαίου. Αλλά γενικώ, μπράβο Βίκη και ευχαριστούμε για την έκθεσή σου. Στάλερ. Ευχαριστούμε κύριε Γκυρό. Η κυρία Κραπίνη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τη Δίκη και τους σκιώδεις ναι. εισηγητές. Αυτός ο κανονισμός θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι ύψης της ε, σημασίας, αλλά Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως ε, αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, για, τον, ε, για τα μέσα ατομικής προστασίας έχει μεγάλη σημασία για, τις, για τα διακοσμητικά στοιχεία ή για τις ελωρίδες που φωσφορίζουν πάνω στα ρούχα, το παράδειγμα που μας έδωσε η Βίκη, πρέπει να ξέρουμε ότι για τον, τα μέσα ατομικής προστασίας, όταν προσδιορίζουμε το πεδίο εφαρμογής, θα πρέπει να αποκλειστούν τα διακοσμητικά στοιχεία αυτές οι φωσφορίζωσες λωρίδες ε, που είναι στα ε, μπουφάν των παιδιών παραδείγματο χάρη δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο στόχος τους είναι να, ε, η ασφάλεια των παιδιών φυσικά μπορεί να συμβάλλει και αυτό όμως εάν δεν προσέξουν και τρέξουν και γίνει δυστύχημα δεν πρόκειται να αποτρέψει το δυστύχημα η φωσφορίζωσα λωρίδα πάνω στα ρούχα. Ε, οι σε αυτές λωρίδες ε, στα μπουφάν δεν προστατεύουν, ξαναλέω, κανέναν ε, εάν γίνει δυστύχημα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα ε, στα είδη που ε, μπορεί να συμβάλλουν στην ασφάλεια αλλά δεν την κατοχυρώνουν. Σε σχέση με την περίοδο εγκυρότητας. Ε, ίσως χρειάζεται μια ελάχιστη τέτοια περίοδος ισχύω ε, για την ε, πιστοποίηση των ειδών αυτών, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Thank you, Mrs. Σας ευχαριστούμε κυρία ε, η κυρία Φόρντ ε, θέλετε να απαντήσετε ή να ακούσουμε την Επιτροπή. Εκτός μικροφώνου λέει η κυρία Φόρντ καλύτερα να ακούσουμε την Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε. Εκτός μικροφώνου επίση. Σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνατε και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ως προς το πεδίο εφαρμογής, ξέρετε ότι για τις ε, ε, συμβαστικές τροπολογίες 1 και 2 ε, ο Επίτροπος πρότεινε την της του αποκλεισμού των γαντιών για ιδιωτική χρήση. Όπως σας είπαμε, Πέραν αυτού θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες που κάνετε για να βρεθεί μια κοινή λύση από τους συνομοθέτες. Για τη συμβαστική τροπολογία για σε τα φωσφορίζοντα τμήματα ρουχισμού, Συμφωνούμε ότι είναι ευπρόσδεκτη η τροπολογία για την ε, παρατεταμένη επαφή με το νερό. Θα ήθελα τώρα να κάνω μια παρατήρηση ίσων σημασίας για τη διατύπωση που σχετίζεται με την συμβαστική τροπολογία 3 και κυρίως ε, την 7-5α παράγραφο όπου αναφέρεται ότι θα μπορούσαν ε, τα πιστοποιητικά να ανανεωθούν αυτόματα και ότι δεν υπάρχει διαδικασία για αυτόματη ανανέωση. Το επίρρημα αυτόματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται μέσα σε αυτή την παράγραφο και ε, καλύτερα να παραλυθεί. Η συγγήτρια. Μπορείτε να μου το ξαναπείτε αυτό. Πού είναι αυτό το automatically, το αυτόματα. Είναι στην παράγραφο από το 5 α η τρίτη παράγραφος από το τέλος. Λέει, όταν ο οργανισμός κοινοποίησης έχει επιβεβαιώσει ότι καμία αλλαγή μπλα μπλα μπλα και ο οργανισμός ε, κοινοποίησης πρέπει αυτόματα να ανανεώσει το, το πιστοποιητικό. Το αυτόματα, η λέξη αυτόματα περιπλέκει τη διατύπωση. Καταλαβαίνω, ναι, ναι, όντως μάλλον είναι περιττό. Θα ήθελα τάχει να επανέλθω σε κάποιες εξαιρετικές παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Πρώτον, για το άρθρο 17 και την τροπολογία που προτείνει διαγραφή του άρθρου 17 λέει ότι θα πρέπει να ταξινομηθούν τα μέσα ατομικής προστασία κατηγορίες που προβλέπονται στο παράρτημα 1 και η Επιτροπή αν κατάλαβα καλά μα ζητά να το διαγράψουμε αυτό και το αναφέρουμε αλλού. Αν το έλεγχο έχει πρόβλημα δεν έχω πρόβλημα, Απλώ πείτε το μας. Είναι γλωσσικό το ζήτημα, διότι ούτω ή άλλω παραπέμπουμε στα παραδείγματα αλλού, στο διατακτικό. Δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα. Για τα, τις ανώτατες ε, και ε, ελάχιστες προθεσμίες ε, τουλάχιστον πέντε χρόνια ή τα πιστοποιητικά λίγουν εκ νέων σε μια περίοδο μέχρι πέντε χρόνια. Ας γεφυρώσουμε το χάσμα. Κάποιοι λένε πρέπει να είναι το ανώτατο όριο, κάποιοι λένε το ελάχιστο τα πέντε χρόνια. Μήπως να προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. κατά το όριο 7 και κατελάχιστο κάτι άλλο. Μπορεί ένα-δύο χρόνια να είναι προσφορότερο εάν είναι ένας τομέας όπου η τεχνολογία είναι τέτοια, ε, ανανεώνονται πολύ γρήγορα τα ίδια. Ε. θα καταθέσουμε μια συμβαστική με δυο τρεις αναλλακτικέ και το ξανασυζητάμε στον τριμερή. Αλλά νομίζω ότι πλησιάζουμε τη λύση. Για τη, τα κράνη μοτοσυκλέτας, βεβαίως, είναι ένα μέσο ατομικής προστασίας ναι. ε, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποια που προβλέπονται και σε άλλα νομοθετήματα. Πάντω, εγώ, την, κύριε Ρόσφο, να την υπερψηφίσω αυτή την τροπολογία. Α, για τα μπουφάν, λέγατε, όχι μόνο για τα κράνη και τα μπουφάν μοτοσυκλέτες, μάλιστα. Και τα δύο, και τα δύο, όχι το ένα ή το άλλο, και τα δύο. Υπενθυμίζω ότι ο στόχος είναι να απλουστεύσουμε την υφιστάμενη διαδικασία για να αναγνωρίζουμε ευκολότερα τους οικονομικούς φορείς στην αλυσίδα αξίας, αν κάτι πάει στραβά. Η υφιστάμενη για τα μέσα ατομικής προστασίας υπάρχει εδώ και 25 χρόνια. Έχουν αποκλειστεί τα γάντια οικιακής χρήσης. Ε, το τελευταίο τέταρτο αιώνα και κανείς δεν παραπονέθηκε γι' αυτό. Και, αλλά ήταν νομικά ασαφές να κατάλαβα. Καλό να το διασαφίσουμε λοιπόν και να πούμε α, άμα σας προστατεύουν από τη θερμότητα τα γάντια να πρέπει, θα πρέπει να τα ε, θεωρούμε ως μέσα ατομικής ε, προστασίας. Ακούω αυτά που μου λέτε και θα τα λάβω υπόψη. Ελπίζω να υπάρξει η πλειοψηφία για να διευκρινίσουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα στον τριμερή. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε και ε, σας επιστρέφω το θόκο. The next file is the um, opinion. Επόμενο θέμα, Γιάννης Νίλσον, γνωμοδότηση για τη διάδοση ε, στοιχείων απαρατήρησης από δορυφόρο για εμπορικούς σκόπους. Α, όχι. Διορθώνει η Πρόεδρος, έχασα τη σελίδα μου και δεν σας τα είπα καλά. Ε, δεν είναι αυτό το επόμενο θέμα ακριβώς, αλλά, γιατί είναι το 7 ο αντίκτυπο που έχουν οι εξελίξει στι ευρωπαϊκές αμυντικέ αγορές, στι δυνατότητες ασφάλειας και άμυνα στην Ευρώπη. Σα θυμίζω ότι η Επιτροπή μα γνωμοδοτεί μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις σε αυτό το τομέα και όχι φυσικά καταλαβαίνετε για την αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Έλντικο Γκαλπέλτς που είναι και η συγγήτρια ε, της Επιτροπής μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση και θα μιλήσω και ογκρικά. Με πολύ μεγάλη χαρά είδα ότι έχετε καταθέσει τόσες πολλές τροπολογίες, 76 παρακαλώ, ε, οι συνάδελφοι. Ε, οι περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές εμπλουτίζουν την αρχική πρόταση, τη δική μου και είναι εξαιρετικές θα έλεγα οι τροπολογίες αυτές. Επίσης, με χαρά διαπιστώνω ότι συμφωνούμε με τους περισσότερους συναδέλφους και είδα να συμφωνούν οι συνάδελφοί μου ε, που έκαναν τροπολογίες ε, για την αλλαγή των προτεραιοτήτων. Χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό. Μέχρι τώρα έχουν γίνει απόπειρε να ενοποιηθεί η ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βάγισαν όλε. Είναι ακόμα κατακαιρματισμένη η ζήτηση στην αμυντική ε, αγορά, στις προμήθειες ε, εξοπλισμών και ε, δεν μας βοήθησε και ένα επιπλέον γεγονός τα σχέδια για την ανάπτυξη δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας δεν επέτυχαν ούτε αυτά ουσιαστικά. Οπότε, όταν αρχίσει η ε, αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και του Αλόγου Οργανισμού, θα πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στο σχεδιασμό για προμήθειες αμυντικού υλικού από τα κράτη-μέλη. Αλλιώς δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Γνωρίζω βέβαια ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά και πολλή δρόμος ακόμα. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να ιεραρχήσουμε κάπως τις προτεραιότητές μας. Και αυτές είναι οι διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών ε, και ανήκουν και στη δική μας αρμοδιότητα, ΙΜΚΟ. Νομίζω ε, ότι είναι αρκετά καλές οι ε, τροπολογίες. Πολλοί συνάδελφοι είναι ειδικοί στο θέμα και έχουν κάνει πολλές τροπολογίες. Λοιπόν, ε, συμφωνώ με τους σκιώδεις των σοσιαλιστών, φιλελευθέρων, πρασίνων και συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. συμφωνώ απολύτως εκεί που λέγουν ότι Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν την οδηγία υπαριθμών 81 του 2009 στην εθνική τους νομοθεσία, οπωσδήποτε, και να την ε, υλοποιούν ε, πλήρως και απολύτως, έτσι ώστε οι εξαιρέσεις να περιορίζονται στο ελάχιστο και να μειώνεται έτσι αυτός ο κατακαιρματισμός των διαφόρων κανόνων και η πανσπερμία κανόνων που έχουμε για τις ε, δημόσιες προμήθειες. Σας εφιστώ την προσοχή στο άρθρο 346 για τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ορίζονται οι εξαιρέσεις. Αυτές θα πρέπει ε, να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχει από χρόνο λόγος ε, στην πράξη και ουσιαστικό δηλαδή. Ε, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της έτσι ώστε να δημιουργηθούν ίσοι κανόνες και προϋποθέσεις στην αγορά της αμυντικής βιομηχανίας και να σταματήσουν οι πρακτικές τρέβλωσης της αγοράς. Είπαμε, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτω απαραίτητο, πρέπει να σας πω ότι προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα τις τροπολογίες των συναδέλφων να αναφέρουν ε, ε, τους νέους τρόπους ε, προκήρυξης διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις. Είναι πολλές αυτές οι τροπολογίες και είναι και ένας από τους τομείς όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και να επιτύχουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτές τις νέες δυνατότητες. Τι εννοώ εδώ. Διάφορα κριτήρια για ομαδοποίηση των προμηθειών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι μακρύς ο κατάλογος των στοιχείων αυτών που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε. Ε, είναι αρκετά εύγλωτα τα παραδείγματα. Αυτός ο νέος τρόπος δηλαδή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και άλλων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος και το οικονομικό και το διοικητικό και ε, τις ε, της αγοράς. και θα πρέπει σιγά σιγά να καταργηθούν, ε, σταδιακά εννοείται, αυτές οι διαφορές και αυτές οι στρεβλώσεις στην αγορά. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που θα θέλαμε να συμμετέχουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, τεχνολογική και βιομηχανική, να ολοκληρώνονται ε, με άλλο τρόπο οι ε, διαγωνισμοί, ε, με άλλο τρόπο και όχι με αντισταθμιστικά ωφέλη, τα περίφημα offsets, για να σταματήσει ο σημερινός κατακαιρματισμός. Βέβαια ξέρω ότι υπάρχουν και κυβερνήσεις που διαφωνούν και μεταξύ αυτών είναι και η δική μου κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις έχουν δικές τους προτεραιότητες και θέλουν να ευνοήσουν τη δική τους αμυντική βιομηχανία για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να τονώσουν τις δικές τους επενδύσεις. Αυτό είναι προφανές και ε, κατανοητό. Αλλά η καλή συνεργασία σημαίνει και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Ε, ε, και εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει αυτό να το υποστηρίξουμε. Και ταυτόχρονα να προστατεύουμε πάντα το απόρριτο των πληροφοριών. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν και τα κράτη-μέλη και εμείς οι ίδιοι ότι Υπάρχει μια αλληλεξάρτηση στην Ευρώπη και ακριβώς αυτή είναι μια κατεξοχήν ε, βιομηχανία που ε, φαίνεται ε, πάρα πολύ αυτή η αλληλεξάρτηση. Ξέρω ότι το νόμισμα έχει δύο πλευρές και βλέπω να το αναφέρεται αυτό και στις ε, τροπολογίες σας. Είναι δύσκολο να παντρέψουμε τις δύο πραγματικότητες. Ε, προσπαθήστε, συνάδελφοι, να βάλετε λίγο στην άκρη τις προσωπικές σας πεπιθήσεις και τα εθνικά σας συμφέροντα, διότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα είναι μια γνωμοδότηση ως Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, και να βελτιώσουμε τις δυνατότητες αυτού του κλάδου μέσω και μακροπρόθεσμα. Δεν έχει νόημα τώρα να συνεχίζεται αυτό ο κατακαιρματισμός των αγορών. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους συναδέλφους, αν γίνεται, να υποστηρίξετε τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες για να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση κάπως συνεκτική και η οποία να αντανακλά τις κοινέ μας θέσεις και τις κοινέ μας σκέψεις και τους κοινού μας στόχους. Ευχαριστώ πολύ. I don't think any of the shadows are present, um, but Catherine Steiner is going to speak. Η κυρία Στάιλερ θα μιλήσει για λογαριασμό του Σέρχιου Γκουτσιέρες. Thank you. I'm, I'm, I'm, uh, the, the, the rapporteur gives the... Σας ευχαριστώ κύριε Στάιλερ. Να τον συμπαθάτε λίγο πιο εισηγητής. Δεν μπόρεσε να παραστεί αλλά μου είπε για λογαριασμό ότι να σας πω τα εξής, να σας διαβάσω από ένα σημείο το οποίο μου έδωσε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την καλή της γνωμοδότηση, για τη συνεργασία της. Τα περισσότερα που ήθελαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες έχουν καλυφθεί και από τη δέσμη των ε, συμβαστικών. Επίσης θεωρούμε ότι στην πρώτη τροπολογία καλύτερα που θέλαμε, ε, παρόλα αυτά όμως λέμε ότι θα πρέπει να να λάβουν υπόψη ε, όσα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2013. Αυτά δεν ήταν απόψη για διάφορους εμπλεκομένους της ε, ΚΕΠΑ. Και ε, αυτό αφορά και την, ε, το πολύπαριθμόν 3. Όμως, καλύτερο το πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία κρατών μελών, να μην έχουμε επικάλυψη ενεργειών και επίσης υπάρχουν έμεσες συνέπειες σε διάφορους αλληλοεπηρεαζόμενους τομείς, οπότε να έχουμε μια ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Κατόπιν έχουμε τις συμβαστικές 5 και 6 και θεωρούμε ότι εκεί είναι θετικό, ότι αναφέρονται οι ΜΜΕ, πάρα πολύ θετικό αυτό, ακριβώς όπως τα είπε και η συγγήτρια. Ε, και έχουμε διάφορα σημεία που η πολιτική μας ομάδα ε, συζήτησε και δεν καλύπτονται από τη δέσμη των συμβαστικών. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικά σημεία και θα θέλαμε να μας υποστηρίξετε. Πρώτα-πρώτα είναι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, τις περικοπές στον προπολογισμό άμεσα περισσότερες χώρες, γιατί έτσι η άμυνα δεν μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία της. Να ε, χρειάζεται συντονισμό όσον αφορά την ε, ΚΕΠΑ, να μην έχουμε επικάλυψη ενεργειών και επίσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία των προτάσεων του 2009 για κάποια κέντρα εξάσκησης όσο προβλέπονται στον κανονισμό την οδηγία 2009, τη 43 και την 81 και να μπορούν να οι ΜΜΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις συμβάσεις που αφορούν την άμυνα. Αυτά έχει ζητήσει ο σχεδόν ηγητής των σοσιαλιστών να τονιστούν περισσότερο. Εξυγχρονισμός πάλι των συμβάσεων και διαγωνισμών προμηθειών. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τις ηλεκτρονικές προμήθειες. Και έχουμε σχετικά για την ε, τροπολογία 72. Σα ευχαριστούμε συγγήτρια και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν έσει ο τέλο οι διαπραγματεύσει για τι τροπολογίε. Κάποιο άλλο θέλει να μιλήσει για τους χιώδες. Ντάντον. Εκ μέρου του θέλω να σας πω που είναι ο σχεδοσυγητής για μα. δεν μπορεί να παραστεί αυτό. Οπότε πρώτα πρώτα θα ήθελε να ευχαριστήσει και την συγκεντρική και τους σχεδοσυγητές για τη συνεργασία τους και για τη συνεργασία για ένα τόσο σημαντικό για όλους θέμα Όσον αφορά την τελευταία εκδοχή των συμβαστικών, έχουμε 18, 7 ε, και 8 εντάξει, χωρίς άλλες παρατηρήσεις. Δυστυχώς κάποιες παρατηρήσεις μας δεν καλύφθηκαν. Ευχαριστεί την εισηγήτρια και την γραμματεία γιατί κάλυψαν αυτά που ζητήσαμε στο 4 και ως προσθήκη δέχτηκε το, την τροπολογία 29, τη συμβαστική 5. Ο κ. Γιάκεβιτς είναι λίγο απογοητευμένος ως προς αυτό το σημείο για να ληφθούν υπόψη οι διακομματικές απόψεις για τις ΜΜΕ. Δυστυχώς όμως η τροπολογία του υπαριθμού 38 βγήκε από τον συμβασμό. Και ο Γιάκεβιτς επίσης θεωρεί θετικό το, το πρώτο σχέδιο κειμένου για την ε, συμβαστική. Οπότε, εάν δεν καλύψετε την τροπολογία μας, λέει ότι δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Τα ρυθμιστικά πάρα πολύ σημαντικά και λέει ότι αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί μακρόπνο μόνο όταν σταματήσουν να υπάρχουν ε, στοιχεία στάθεια στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Για την ECR πάντω και η συμβαστική 5 είναι κόκκινη γραμμή. Δεν έχει πολλά να πει για τις υπόλοιπες συμβαστικές, απλώς τώρα για το 2 και για το 6 το... πρόκειται να σας πει ποια είναι η απόψή μας, αλλά καταλαβαίνουμε και θα συμβαστούμε το ότι θα ε, ψηφίσουν οι άλλε πολιτικέ ομάδε. Θα ζητήσουμε από τη γραμματεία χωριστή ψηφορία. Πάση περιπτώσει αυτά θα τα πούμε στην εισηγήτρια με email. Αυτά εκ μέρου του κυρίου Γιάκεβιτς. Τώρα κάποιε προσωπικέ μου παρατηρήσεις γιατί είμαι για το ισχυρό συντονιστή. Εγώ είχα προβληματιστεί για το που πάει αυτή η υπόθεση. Και θεώρησα ότι τώρα εξευρωπαίζουμε ε, τις προμήθειες της αμυντικές και θεώρησα ότι αυτό δεν είναι τόσο σόφρον λύση να υπάρχει ένα καθεστώς που να διέπει τις ε, προμήθειες και αυτό να κάνουμε. Ή πρόεδρος. Για τους ελευθέρους θέλει κανείς το λόγο. Για την αριστερά, για τους πράσινους. Καλώς. Μπορεί να δευτερολογήσει τώρα η συγκίτρια. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές και τους συντηρητικούς για τα σχόλιά τους. Είναι γεγονός. Δεν μπορούν όλες οι τροπολογίες να συμπεριληφθούν στις ε, συμβιβαστικές. Θα πρέπει να έχουμε τον ίδιο κοινό στόχο, να μην αλλοιώνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διατηρήσουμε το στόχο μας στις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν μπορούν να μπουν όλες οι τροπολογίες. Ο Σέρχιο Γκουτιέρες κάνει λόγο για την οικονομική κρίση που σήμαινε και περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Και μιλάει για την τροπολογία 72. Αυτή συμπεριλαμβάνεται τώρα στο συμβιβασμό. Και αυτό μπορεί εύκολα να διευκρινιστεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει μεγάλη σημασία να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμφωνώ. Και σε ό,τι αφορά τα σχόλια των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και του συντονιστή τους, είναι γεγονός ότι τα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι κόκκινη γραμμή ε, για να εγκριθεί αυτός ο συμβιβασμός, αλλά πρέπει να σας πω ξεκάθαρα ότι αυτή η πρακτική των offsets όπως λέγεται είναι περίπλοκη, ασαφής, θολή και σκοτεινή. Και αυτό δεν βοηθάει ε, στο να ενοποιηθεί αυτή η κατακαιρματισμένη αγορά που πρέπει οπωσδήποτε γιατί είναι τεράστιες οι δαπάνες, ε, οι αμυντικές, χωρίς απαραίτητα να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Χρειάζεται συντονισμός Συντονισμός δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε όλοι ένα το ίδιο, ε, σημαίνει ότι θα σχεδιάζουμε, θα συντονιζόμαστε, θα ξέρουμε τι δαπάνες σχεδιάζει η κάθε χώρα στην αμυντική της ε, ε, προμήθεια. Αυτό είναι καλό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλιώς θα έχουμε άχρηστες δαπάνες. Το ξέρω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε παράλληλες γραμμές, αλλά είναι σημαντικό να χρηματοδοτούμε ε, κάτι σε κάποιο κράτος μέλος ε, και να γίνεται αυτό με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις για να υπάρχει διαφάνεια. Συμφωνώ ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες που ε, έχουν πληγεί λόγω της κατάργησης των αντισταθμιστικών ωφελών που θα πρέπει όμως να βρουν έναν τρόπο να τα αντισταθμίσουν την έξι συμβιβαστική τροπολογία δεν συμφωνώ με το όσα είπατε. Ο κύριος Γιακέβης δηλαδή, ε, συμπεριλαμβάνονται τα σχόλιά του, τον έχω υποστηρίξει. Εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό διμερός για να το ξεκαθαρίσουμε. Λυπάμαι που οι συντηρητικοί και οι μεταρρυθμιστές δεν υποστηρίζουν αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί πιστεύω ότι θα άξιζε και θα μπορούσε να είναι κοινή η γνωμοδότηση όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank Η κυρία Χαράνσοβα, ε, συγγνώμη που άργησα, αλλά είχε πολλή κίνηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγητρία, διότι προσπάθησε να λάβει υπόψη αποκλίνουσες απόψεις ε, για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι από πολλές πλευρές είναι ευαίσθητο αυτό το ζήτημα για πολλά κράτη-μέλη, ε, κυρίως ε, σε, σε κράτη όπου υπάρχουν προμηθευτές αμυντικού εξοπλισμού και θα ήθελα να το λάβετε και αυτό υπόψη. Για την παράγραφο 5 υπάρχει αυτό το θέμα των offsets. Ίσως δεν είναι το καλύτερο σύστημα, αλλά χρειάζεται μια εναλλακτική λύση, τουλάχιστον για τα μικρά κράτη-μέλη. Ε, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η, το σταδιακό, η σταδιακή απάλληψη των offsets χωρίς μια ε, εναλλακτική λύση θα είναι επιζήμια για την οικονομική κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, επίσης οι διατάξεις ε, του άρθρου 21 της Οδηγίας 81 για την υπεργολαβία λειτουργούν σαν αντιστάθμισμα των αντισταθμιστικών. Ε, όμως, προσοχή γιατί διοικητικά είναι περίπλοκο. Τα κράτη-μέλη ισχυρίζονται ότι σε περιπτώσεις όπου ε, είναι εφαρμοστές οι διατάξεις για την υπεργολαβία, τότε ε, είναι μεγαλύτερο το κόστος και χρειάζεται και περισσότερος χρόνος ε, για τις προμήθειες. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο άχθος και για τους υπεργολάβους και δεν ξέρω αν είναι προετοιμασμένοι δεν υπάρχουν ικανοποιητικές λύσεις, σύντομα δεν θα έχουμε offsets ε, αφενός και αφετέρου δεν θα έχουμε κάτι που να τα αντικαθιστά. Άρα δεν θα είναι εξισορροπημένη η αμυντική αγορά στην Ευρώπη. Ελπίζω να τα λάβετε υπόψη αυτά και να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Ζητώ αναδιατύπωση της τροπολογίας 5 ήδη. Ελπίζω επίσης πως ε, θα κάνει κάποια βήματα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής ε, για να ε, βρει ένα καλύτερο τόπο να συνδέσει τον τομέα της άμυνας με άλλους βιομηχανικούς τομείς και ζητώ κλείνοντας συγγνώμη και πάλι που άργησα με την κίνηση που είχε. Σας ευχαριστούμε. Επόμενο σημείο. διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. Ε, είναι σχέδιο οδηγίας. Η Επιτροπή Βιομηχανίας είναι η καθήλυνα αρμόδια. Από την ομάδα μας ο Γένς Νίλσεν ε, είναι ο εισηγητής μας και έχει δώσει το σημειωματάκι στην Κάθριν Στάιλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Έχω το σημείωμα του Γένση και θα σας τα διαβάσω. Ζητά συγγνώμη πρώτα απ' όλα, διότι είναι σε μια υπουργική συνάντηση στη Στοκχόλμη, γι' αυτό δεν ήρθε. Ο τομέας αυτός γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκοσμίω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε η διαστημική αγορά για τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται ότι παρακολύεται από την απουσία ενός συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου στην Ευρώπη, προτινόμενο οδηγεί για τη διάδοση δορυφορικών, γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, έχει ως στόχο να ρυθμίσει την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι χρειάζεται κοινή νομοθεσία για να κυκλοφορούν ελεύθερα τα, δεδομένα, τα δορυφορικά δεδομένα, να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς και τους παρόχους. Ταυτόχρονα λοιπόν αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίε για την ασφάλεια αλλά και τα εθνικά συμφέροντα είναι πάρα πολύ δύσκολη εξορρόπηση αυτών των δύο διότι μπορεί να είναι διτής χρήση τα δορυφορικά δεδομένα στρατιωτική και μη χρήση. δηλαδή ο εισηγητή πιστεύει ότι ε, έχει, ε, ε, είναι αξιοποιήσιμη η οδηγία στον διαστημικό τομέα ο στόχος είναι να επεξεργαστούμε επικοδομητικά το σχέδιο οδηγίας, ούτως ώστε να έχουμε συμφωνία με συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εμπλεκόμενους φορείς. Ε, ο εισηγητής και οι σχεδόντες έχουν κάνει τη διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς. Ο στόχος είναι να υπάρξει συγκροτηθεί μια ενιαία αγορά για αυτά τα δορυφορικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, όμως σε σχέση με το περιεχόμενο σχεδίου οδηγίας φαίνεται ότι γίνεται μια κάπως διαφορετική αποτίμηση της κατάστασης και γι' αυτό ο συντάκτης ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ήδη υποβάλει ένα έγγραφο εργασίας που μοιράσαμε στα μέλη της Επιτροπής ΙΜΚΟ όπου τονίζεται τα βασικά σημεία που χρειάζονται για την ευκοδομητική επεξεργασία του σχεδίου οδηγία ε, και ε, προτείνονται διάφορε βελτιώσει. Θα ήθελα εν συντομή να αναφερθώ σε κάποια από αυτά τα σημεία που θα ήθελε οι εισηγητή να βελτιωθούν. Είναι τα εξή. Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι υπάρχουν ελλείψει στην προπαρασκευαστική φάση, παραδείγματο χάρη το πρόβλημα με τους ορισμούς, τα πιστήρια, η αξιολόγηση αντικτύπου είναι ποιοτική τική και δεν γίνεται επαρκή ε, εξεργασία των δεδομένων κόστους ωφέλους. Επίσης ε, δεν ε, εξετάζεται διεξοδικά το νομικό μέσο που προτείνεται. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο ποια κολλήματα υπάρχουν στην ενιαία αγορά και πώς ακριβώς μπορεί αποτελεσματικά να αναβαθμιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι υποχρεώσεις για την ε, αναλυτική εξέταση και για την πιστοποίηση θα οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος. Ε, ο στόχος της οδηγίας θα πρέπει να υπάρξει μια νέα χώρα για την, διάδοση αυτών των δεδομένων, να τον προωθηθεί η καινοτομία και η νέα τεχνολογία και να υπάρξει ένα θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς όπως η γεωργία, το λιανικό εμπόριο, η χωροταξία, ο σχεδιασμός των μεταφορών, ε, πετρελαϊκή η βιομηχανία και ούτω καθεστής και ούτω καθεξής. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτή την πρόταση ε, για να υλοποιηθούν οι ε, προτινόμενες βελτιώσεις θα πρέπει να υπάρξει καινοτομία και το, κυρίως αυτό ισχύει για τη διάδοση των γεροσκοπικών δεδομένων. Φυσικά θα πρέπει να ε, μην τίθεται ζήτημα εθνική ασφάλεια και όπω βλέπουμε και από την εμπειρία των ΗΠΑ υπάρχουν ε, σοβαρά στρατηγικά συμφέροντα που σχετίζονται με τη διεύρυνση αυτού του τομέα δορυφωνικών ε, δεδομένων και πλήττεται ολόκληρη βιομηχανία. Θα πρέπει να ληφθεί και αυτό η υπόψη. Η διάδοση δεδομένων υψηλή αυκρίνης από τρίτε χωρίς είναι άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μα εξηγήσει πώ ακριβώ θα αποφύγουμε στρεβλώσει μέσα στην ενιαία χώρα που θα οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσει για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σα ευχαριστούμε που ακούσατε αυτές τις παρατηρήσεις και σίγουρα ο εισηγητή Γιάννης Νίλσεν θα ε, θεωρήσει ότι είναι ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε σχόλια και παρατηρήσει έχετε να κάνετε. For e uh, Ο Τόελκ, ο Λάμπερτ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για την καταπληκτική παρουσίαση του μηνύματος. Ε, έχω λίγο τις επιφυλάξεις μου και τις αμφιβολίες μου για το περιεχόμενο. Πάντως η παρουσίαση ήταν εξαιρετική. Γιατί τα λέω αυτά, θυμάμαι καλά. Ήταν από τις προτάσεις που ήταν στο Refit. Και τώρα το βγάλανε και από την Επιτροπή μας και επί της ουσίας είναι αρμόδια Επιτροπή Οβιομηχανίας, η Ήτρε, και εμεί είπαμε να μελετήσουμε τα 10 πράγματα και όλο αμφισβητούμε, αμφιβάλλουμε κτλ. Τώρα πού βρισκόμαστε. Μέσα στην αμφιβολία είμαστε. Αν θέλει η Επιτροπή μας να επεκταθεί στην εσωτερική αγορά, εκεί θα πρέπει και να παραμείνουμε. Αν γνωρίζουμε ότι αλλάζει η αγορά, θα πρέπει να το πούμε. Και αν κάποιες χώρες, έξι ας πούμε, ακολουθούν το δρόμο τους, να το πούμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι είπα, στραβάρμενίζουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τους ενεχομένους και τα λοιπά. Δηλαδή, μαθαίνουμε περισσότερα, ξέρουμε περισσότερα και κάνουμε λιγότερα. Ε, δεν μπορεί να καταλήξει και η συζήτησή μας, δεν επιτρέπεται. Τι λέει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ότι έχουμε αρκετούς λόγους έτσι ώστε σε πρώιμο στάδιο να επέμβουμε για να φτιάξουμε κανονισμούς και να φέρουμε προτάσεις και να μην το ξαναστείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το μελετάει ακόμα ένα χρόνο. Μπορώ να σας πω τι θα κάνει μετά από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ξέρει περισσότερα και θα κάνει λιγότερα. Το μήνυμα λοιπόν θα μπορούσε να είναι και περιμένω από τους συγητές εγώ να έρθουν ε, με πιο στεναρά στοιχεία και να ζητήσει υποστήριξη. Να πούμε θέλουμε ένα τέτοιο κανονισμό, θέλουμε να πάμε προς την κατεύθυνση αυτή, ναι ιού. Όχι, δεν είναι κανονισμός, διορθώνει ο μιλητής, είναι οδηγία, λέει ο κύριος Βανίστεροι. Λοιπόν, αυτό το δρόμο θέλουμε να ε, διαλέξουμε. Αν ναι, να δούμε και μέχρι πού θα πάμε. Αλλά το πλαίσιο κανονικά θα πρέπει να είναι σαφές. και να υπάρχει και ένα οικονομικό αποτέλεσμα αρκετό που δεν έχουμε σήμερα. Ε, πρόκειται για τα στοιχεία, για τα big data, τα δεδομένα που είναι κρίσιμα και δεν ξέρουμε ε, καν αν θα χρησιμοποιούνται μετά από 10 χρόνια και αν συσσωρεύονται ε, τα δεδομένα που θα καταλήξουμε. Παρακαλώ λοιπόν να επιταχύνουμε. Ακούγοντα και ε, την εισηγήτρια και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Σκιώδη, έχω την αίσθηση ότι συμφωνούμε όλοι ότι η σημερινή εκδοχή της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αρκετές ελλείψεις και σοβαρές. Μπορεί να διαφωνούμε ως προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά συμφωνούμε στη διάγνωση. Εγώ δεν έχω πιστεί από τη λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πρόταση αυτή όπως έχει διατυπωθεί ή όπως την έχουν συλλάβει θα επηρεάσει θετικά την αγορά. Ούτε είμαι καθόλου βέβαια ότι θα αυξήσει την ευημερία, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. Επίσης δεν έχω πιστεί καθόλου ότι θα βοηθήσει στην προστασία της ιδιωτική σφαίρας των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλειά τους. Για παράδειγμα, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν ότι μόνο υψηλή ευκρίνεια γεωσκοπικά δεδομένα είναι ευαίσθητα. Αυτό είναι ξεπερασμένη άποψη. Μπορεί και με κανονική ευκρίνεια εικόνες και στοιχεία ε, να έχουν ζητήματα προστασία και ιδιωτικότητα. Ποια είναι η ευρωπαϊκή λύση όμως και η προσέγγιση. Η ευρωπαϊκή δορυφορική βιομηχανία είναι από τις μεγάλες μας επιτυχίες στην αγορά η αύξηση της ζήτησης ε, για τις υπηρεσίες ε, τηλεπικοινωνιών είναι θεματική και αναπτύσσεται ο κλάδος ε, με τους καλύτερους ρυθμούς. Είναι από τους καλύτερους και τους πιο γρήγορους. Δηλαδή να προσέξουμε στην νομοθεσία μήπως όταν την εγκρίνουμε, μέχρι να την εγκρίνουμε, μήπως έχει καταστεί και αυτή απαρχιωμένη και δεν βοηθάει καθόλου τον κλάδο θα πρέπει να δούμε τι προστατεύουμε. Κάποια δεδομένα και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με ζητήματα ασφαλείας, καλώς. Αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαια ότι αυτή η πρόταση καθιωδήποτε τρόπο επιτυγχάνει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμφωνώ πολύ με την εισηγητρία προς τις ε, αδυναμίες της πρότασης. Εγώ θυμάμαι όταν είχε έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ανταλλαγή Απόψεων, το είπαμε και είπα ότι ε, πρόκειται μόνο για εμπορικούς ε, χρήστε, ότι δεν καλύπτει το Γαλιλαίο και αυτό μου είχε φανεί περίεργο τότε. Ε, και είναι πολύ λίγες οι χώρες εκείνες που έχουν δορυφόρου και παράγουν τέτοιου είδους εμπορικά δεδομένα. Πρέπει να προβληματιστούμε πολύ, να το ξανασκεφτούμε πώς πρέπει να το αναπέμψουμε να το ξανακοιτάξουν. γιατί η δική μου πολιτική ομάδα ήταν σημαντικό. Οποιαδήποτε νομοθεσία σε αυτό το τομέα δεν θα πρέπει να εγκλωβίζεται σε μια παλιά τεχνολογία και να έχουμε εμπορικό στη συνέχεια μειονέκτημα. Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα καν τα θέματα ασφαλείας και προστασίας. Γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο σε έναν ορισμό του προβλήματος και δεν το βλέπουμε σφαιρικά. Έχουμε πολλή δουλειά φυσικά για αυτά τα προγράμματα, τα, τα προβλήματα συγγνώμη, και θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε. The, um, Δεν είναι εδώ ο Σκιώδης ε, για τους βέτρους η... για, λογαριασμό της ε, Άλτε θα μιλήσει κύριε Χάντζοβε. Ευχαριστώ πρώτα ευχαριστούμε και την εισηγήτρια για την κυρία Στάλερ που μίλησε για λογαριασμό της ηγήτριας, οπότε να σας πω εγώ τι έχει να πει ο Αντώνας, ο οποίος ε, δεν μπορούσε να έρθει αυτός, οπότε ε, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για αυτήν την αγορά δεν έχει ακόμα πιστεί όσον αφορά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται κάποια θέματα που προτείνει να τα εξετάσει. ο λέει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή να προσαγγεί κάποια στοιχεία όσον αφορά τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά ε, σε σχέση με το ότι υπάρχει φραγμό από την έλλειψη σχετική νομοθεσία. Επίση, θα πρέπει να καταστήσει σίγουρο το ότι δεν θα είναι ο κανονισμός αυτός ένας φραγμός για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην παγκόσμια αγορά. Μην έχουμε κάποιους ε, περιορισμούς που αφορούν Φερρυπίν την ασφάλεια. Το θέμα είναι αν θα ε, υπάρχουν κάποιο είδους συστήματα πιστοποίηση με αναλυτικέ εξετάσει, screening, περίπλοκα κλπ. ανεξαρτήτω του τι κάνουν ε, τα, οι, αυτοί οι υπάρχοι στην επικρατεία των κρατών μελών. Επίση, τονίζει ο κ. Γκόγκα ότι αυτά τα δεδομένα υψηλή ευκρίνεια δεν είναι τόσο αξίας όταν έχουν περάσει από την επιστοποίηση. Γι' αυτό και λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαδικασία ταχύτερης παροχής της πιστοποίησης από ό,τι ισχύει σήμερα. Επίσης, θα ήθελε να απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εξηγήσει εκείνη γιατί διάλεξαν ε, αυτή την περίοδο των 70 μερών για την χορήγηση της πιστοποίησης. Είναι αρκετό αυτό το διάστημα να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών. Επίσης, τονίζει ότι είναι ανοιχτό σε συζήτηση και θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω να προσαρμογάγει στοιχεία για το ότι αυτή η πρόταση είναι ή δεν είναι παράδειγμα ευφυούς νομοθεσίας. E ε, δεν βλέπω κανένα σκιώδη από την ΚΟΕ. E. Κανένα από του πρασινου ποιο αλλο θέλει το λόγο. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Βρήκαμε κάποιον. Αγκώστα Γκονζάλες. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για το αν είναι καλό ή όχι για την αγορά είναι μικρή αγορά, αλλά μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό. Ε, η ασφάλεια είναι ένα κόλλημα για την πρόσβαση στα δεδομένα υψηλής ευκρίνειας. Γιατί υψηλής ευκρίνειας, διότι τα ίδια τα κράτη-μέλη έχουν καταλήξει σε αυτά. Ε, ε, εκείνα έχουν τα συστήματα δορυφόρων. Ε, τα δεδομένα χαμηλής ευκρίνειας κυκλοφορούν ελεύθερα. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας, όμως δύσκολα μπορεί κάποιος να παρεμποδίσει την κυκλοφορία ενός πράγματος που ήδη κυκλοφορεί ελεύθερο. Το θέμα είναι τα λεφτά που μπορούν να, να βγάλουν επιχειρήσεις, αυτά θα γίνουν με δεδομένα υψηλής ευκρίνειας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την αγορά ε, λειτουργούν με ίσους ανταγωνισμό, ανταγωνισμού ανεξαρτήτως έδρας. Ε, αυτό είναι ο στόχος της ε, οδηγίας, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη θα πρέπει με μεγαλύτερη ταχύτητα να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα υψηλής ευκρίνειας ε, χωρίς να αποτελούν κόλλημα ε, οι λόγοι ασφαλείας, ε, χωρίς να οδηγεί αυτό σε καθυστερήσει, σε περιττές καθυστερήσεις και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν γκρίζες ζώνες φυσικά και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει κάποιες ε, διευκρινήσεις. Πάντως εμείς κρίνουμε πως σίγουρα θα είναι επωφελής ε, η οδηγία για την αγορά, διότι θα είναι πιο αποτελεσματική, ταχύτερη και ε, ευκολότερη η προσπελασιμότητα των δεδομένων υψηλής ευκρίνειας από πλευράς των κρατών μελών που ελέγχουν τα δορυφορικά συστήματα. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Έχουμε και προθεσμία. Μέχρι τις 12 Μαΐου για τις τροπολογίες 4 Ιουνίου θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Αν η εισηγητής θέλει να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα, είναι δυνατόν αυτό, αλλά θα πρέπει να το δουν οι συντονιστές. Δηλαδή, πώς θα γίνει να ψηφίσουμε στην ΙΦΚΟ πριν την Ήτρε. 22 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη ημερομηνία για την ε, ψηφοφορία ε, στην Ήτρε. Έχουμε εμεί άλλη ημερομηνία στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε στις αρχές. Αλλά από την εμπειρία μου θα έλεγα ότι είναι ε, είναι δύσκολο να καταλήξουμε ε, σε συμβαστικέ τροπολογίε πριν τη συνεδρίαση γιατί είναι η πρώτη εβδομάδα. Τότε έχουμε ημερομηνία μόνο την πρώτη εβδομάδα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. να σα αφήσουμε του συντονιστέ να το συζητήσουμε. τώρα, τώρα, κυρία Στάιλε, συσκευές αερίου. πάνω από 200 τροπολογίες και 4 ε, συμβαστικές τροπολογίες ε, ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Επιτροπή για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους Σκιώδης. Ε, συζητούμε για τις συμβαστικές τροπολογίες, 4 στο αριθμό. Στις 31 Μαρτίου στους ε, συντενιστές τη συζητήσαμε. Έκτοτε κάναμε μια μικρή αλλαγή στην πρώτη συμβαστική Μιλάγαμε για διαρροή συγκεντρώσεων που μπορεί να αποβεί προβληματική και προτείνουμε τώρα για την τροπολογία ένα, διαφορετικό τέλος και σας το διαβάζω. Ε, η διαρροή συγκεντρώσεων όλων των επιβλαβών για την υγεία ε, και για την ασφάλεια ουσιών. Η υπόλοιπη τροπολογία παραμένει ως έχει. Για τις άλλες τρεις θα ήθελα να καταθέσω τώρα δύο προφορικές τροπολογίες. Η μία για το άρθρο 12.9. Θέλω να αλλάξει η διατύπωση και να λέει τα εξής. Οι τεχνικές οδηγίες για αυτό που κάνει την εγκατάσταση και για το σέρβις πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να γίνουν σωστά οι διεργασίες και να είναι ασφαλής η καύση. Ε, και ε, στην εποχή της εγκατάστασης και μετά το σέρβις θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των συσκευών και στην τροπολογία 130 τα ίδια λέμε όχι, διορθώνει η ε, ομιλήτρια το 112 και επίσης 120 εκεί πέρα λέμε για το εμπορικό σήμα και για το ότι αναγράφεται πάνω στην συσκευή και τους σωλήνες Υπάρχουν δύο ξεχωριστές παραγράφους 18.1 και 18.2 για τις συσκευές ε, και για τους σωλήνες, οπότε τώρα προτείνουμε να είναι 18.1. Ε, το σήμα που, αναφέρεται στο παράρτημα 4 θα πρέπει ευανάγνωστα και ορατά να ε, αναφέρονται την, στο πλακίδιο των δεδομένων και στη, στους σωλήνες. Εάν όχι θα πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία και σε ό,τι συνοδεύει ε, τη συσκευή τους σωλήνες. Οπότε γίνεται 18,2 ε, το 18,3 και οι τροπολογίες μας είπε η Ντίτα, νομίζω καλύπτονται από αυτή την τροπολογία και μπορούμε να, καλυφθούμε με τις συμβαστικές τροπολογίες 3 και 4, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που επαναλαμβάνουμε. Ε, παραπέμπουμε στο άρθρο 18 επίσης. Ε, Έχουμε προετοιμάσει και ένα σχέδιο καταλόγου ψηφοφορίας ε, και πρότεινα όσες περισσότερες υπερψήφιση όσων περισσότερων τροπολογιών συναδέλφων μπορούσα και οι 201 έως 205 και 206 είναι από αυτές που δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω διότι θεωρώ ότι εκτίθουν του πεδίου ε, του σχεδίου κανονισμού. Ε, το ίδιο για τη 229 διότι αποδυναμώνει την διατύπωση του σχεδίου κανονισμού. Ζητώ συγγνώμη που τα έμπλεξα τώρα με τους αριθμούς ε, για το 12,9. Πρόκειται για την τροπολογία 29 και όχι για το άρθρο 12,9 την Πέμπτη θα γίνει ψηφοφορία, μία ψηφοφορία για το φάκελο και μία άλλη ψηφοφορία για την ε, διαπραγματευτική εντολή για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να εισέλθουμε στις διαπραγματεύσεις σε τριμερή, δηλαδή με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ και ε, θα ήθελα να ακούσω τώρα τι έχουν να μου πούνε οι um, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνεχίζω τα συγχαρητήρια και τις ε, ε, φιλοφρονήσεις για την παρουσίαση, αλλά τώρα και επί της ουσίας για την πρότασή σας. Εξ ονόματος του κυρίου Μπουσόη, ε, πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με τις συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνούμε. Έχουμε και μια προφορική τροπολογία, θα τη δώσω στην εισηγήτρια. Ε, έχετε πάντως την υποστήριξη του ΕΛΚ σε γενικές γραμμές και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίστερόι είχε μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα επίσκεψη στο Ειτχόβεν της Ολλανδίας, αν θυμάμαι καλά, ε, και πραγματικά θα πρέπει να το κοιτάξουμε γιατί ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία αυτής της αποστολής. Είναι κάτι διαφορετικό και θέλω να σας συγχαρώ γιατί ήταν πολύ ωραία. <laughs> Α επιστρέψουμε στο θέμα μας όμως. Μπράβο, έχετε δίκιο. Πολύ ωραία τα είπατε. Ε, Ντάλτον. Dalton. Εγώ θα είμαι σύντομο. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια που κάλυψε αυτά που θέλαμε στι συμβαστικέ τροπολογίε και με χαρά μας να εγκρίνουμε το κείμενο. Τσάρτζο. Και εγώ να συνεχίζω τους επένου προ την εισηγήτρια Πάρα πολύ ωραίο συμβαστικό κείμενο είναι αυτό στο οποίο καταλήξατε, αλλά μπράβο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βοήθησε. Ιδίω στον αφορά 18. Επ' αυτού είχα κάποιε προτάσει και ήταν πάρα πολύ καλό το ότι τις καλύψανε. Για την ψηφορία τώρα έχω να σας προτείνω κάποιες ιδέες γιατί αυτή η περίπτωση είναι παράδειγμα του πώς κανείς μπορεί να προχωρήσει γρήγορα με, με ψηφοφορίες ομαδικές, πολλών διατάξεων από κοινού. Ευχαριστώ Βίγη. Απλώς να σας πω ότι πρώτα πρώτα ευχαριστούμε για το αξιολογικό κείμενο και συμφωνούμε με όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. Πιο γρήγορα δεν γίνεται, Πρόεδρος. Thank you. Um, commission? Commission? Επιτροπή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να είμαι σύντομο γιατί όλοι είναι σύντομοι πάνω σε αυτά. Όσον αφορά για τι συμβατικέ τροπολογίε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνη Συμφωνία και, αλλά δεν θα ε, σας το έχω ε, σχολιάσει το 129 γιατί σας τα είπε η κυρία Στάιλερ. Α, συγγνώμη για το 229. Γιατί η Ρίκη Στάιλερ τέλο πάντων είπε ότι δεν θα την πρόθεσε. So just like to Στάιλερ, ευχαριστούμε συνάδελφε. Νομίζω ότι προχωρεί η υπόθεση και είναι πάρα πολλές τροπολογίες που έχουν ε, καλυφθεί. Θα τις ψηφίσουμε ώρες μαζί και την Πέμπτη θα γίνει η ψηφοφορία και θα, θα αντιμετωπίσουμε όλο μαζί το θέμα και μετά έτσι θα προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσει μέσω του τριμερούς διαλέγου. Οπότε σα ευχαριστώ όλου και τους σκιώδη. Η γραμματεία όμω μου είπε, λέει πρόεδρος, ότι ο κατάλογο τη ψηφοφορία. θα προβλέπει πολλέ σημαντικές ψηφοφορίε για κάποια θέματα που μπορούν να ψηφίσουν όλα μαζί. Οπότε, γι' αυτό και ελπίζω ότι θα πάει μια χαρά και αποτελεσματικά η ψηφοφορία την Πέμπτη. Πήγα σε μια άλλη επιτροπή, ξέρετε, για μια άλλη ψηφοφορία. Του πήρε 20 λεπτά να, να, να λάβουν θέσει. Και είδα πόσο αποτελεσματικοί είμαστε εμεί στι δικέ ψηφοφορίε. Άρα συνεχίσουμε αυτή μας την παράδοση και ευχαριστώ και την γραμματεία γι' αυτό. Και τώρα, να δούμε τα διάφορα. Τίποτα. Όποτε αρχίσει ε, η συνδύαση των συντονιστών, μόλις έρθουν όλοι εδώ.